Dear colleagues, welcome. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Πάμε στο σημείο 6. Πολύ χαίρομαι λοιπόν που καλωσορίζω εδώ τον καθηγητή Ενρίκο Τζοβανίνη, που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής. Η Επιτροπή μας ενέκρινε τον ορισμό του κύριου Τζοβανίνη στη θέση του Προέδρου τον Οκτώβριο του 2017 και ανέλαβε την 1η Φεβρουαρίου 2018 για τρία χρόνια ο κύριος Τζοβανίνη. Κάθε χρόνο λοιπόν έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον ε, πρόεδρο του ΕΣΚΑΜ, του συμβουλευτικού αυτού φορέα δηλαδή, για να ενημερωνόμαστε για την ε, τελευταία έκθεση πεπραγμένων, η οποία δημοσιεύθηκε για τελευταία φορά πριν από λίγες μέρες και αφορά το 2018. Όπως ε, γνωρίζετε, η έκθεση αυτή αναφέρεται στις στατιστικές προτεραιότητες και μετά το 2020 αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών Δεδομένων επίσης. Και μιλάει επίσης και για το commitment of confidence, για το θέμα της εμπιστευτικότητας των στατιστικών δεδομένων ε, μιλάει επίσης για την βελτίωση δράσεων που έχουν ε, να κάνουν με προηγούμενες συστάσεις του φορέα. Πολλά λοιπόν έχουμε να συζητήσουμε. Την Πέμπτη θα ψηφίσουμε και για το GNI, για το καθάριστο εθνικό εισόδημα. Είναι ένα στατιστικό παζλ και αυτό. είναι κάτι σημαντικό νομοθετικά. Περιμένουμε λοιπόν από τον κύριο Τζοβανίνη πολλά. Έτσι κι ξέρουμε ότι είναι ειδικό στα θέματα στατιστικής, αλλά όχι μόνο. Είναι και πολύ καλός στην εκπόνηση του έργου του για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος. στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να σας τον παρουσιάσω περισσότερο, το γνωρίζετε όλοι. Οπότε σας δίνω και το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους σας. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας για να σας παρουσιάσω την πρώτη έκθεση του Συμβουλευτικού Φορέα μετά την αλλαγή στη σύνθεση γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που ορίστηκα στη θέση του Προέδρου στις αρχές της προηγούμενης χρονιάς, αλλά άλλαξε η σύνθεση του φορέα συνολικά. Και ήταν μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στα άτομα που βέβαια μαθαίνουν όσο περνάει ο χρόνος όλο και περισσότερο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών Δεδομένων είναι πολλές και πολλές από αυτές έχουν να κάνουν βέβαια και με τις επερχόμενες εκλογές. Γιατί μας απασχολεί με ποιο τρόπο τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα δεν ε, ε, διαδίδονται, αλλά σχολιάζονται από τα μέσα ενημέρωσης και ακόμα περισσότερο στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε έχουμε μία ομάδα εργασίας με task force για τα ψεύτικα δεδομένα, τα fake news, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί πολύ περισσότερο στην καταπολέμηση αυτών των ψευδοειδήσεων fake news. Στην έκθεσή μας αναφερόμαστε επίσης και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, Στατιστικών ε, Δεδομένων και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Επιτρέψτε μου να συνοψίσω κάποιες από τις συστάσεις τις ε, οποίες παρουσιάσαμε. Συνολικά είναι 14 οι συστάσεις μας και θέλω να σας πω ότι το 2018 είχαμε και μία έκθεση για την εφαρμογή αυτού που ονομάζεται Commitment on Confidence. Ο στόχος ήταν μια ειδική γνωμοδότηση και τη σύστασή μας τη στείλαμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι στατιστικές υπηρεσίες και, με... και για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή στηρίζει τις δράσεις της Eurostat αλλά όπως ξέρετε το στατιστικό σύστημα είναι ευρύτερο. Περιλαμβάνει τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, αλλά και τις άλλες εθνικές αρχές που ασχολούνται με στατιστικά δεδομένα και που συνεισφέρουν στην δημοσίευση των ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων. Είναι αρμοδιότητα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα, αλλά όπως θα τονίσω και σε λίγο, εντοπίσαμε ένα κενό στο σύστημα και ίσως η Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο θα ήθελε να βρει τρόπο να το αντιμετωπίσει. Λοιπόν, ποιες είναι οι συστάσεις μας. Πρώτα απ' όλα, είναι σαφές ότι με τις μεγάλες και γρήγορες αλλαγές που γίνονται στον οικονομικό, στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα και όχι μάλιστα μόνο στην Ευρώπη, οι ειδικοί για τα στατιστικά δεδομένα έχουν δύσκολη δουλειά να επιτελέσουν, γιατί πρέπει τα στοιχεία τους να είναι ακριβή, να είναι σωστά. Και γι' αυτό ακριβώς η πρώτη μας σύσταση υπογραμμίζει την ανάγκη που υπάρχει στατιστικές υπηρεσίες να είναι πιο δραστήριες, δηλαδή να προλαβαίνουν ε, και να ξέρουν εκ των προτέρων τι είναι αυτό που έχει σημασία να προλαβαίνουν τα γεγονότα και να μην τρέχουν πίσω από αυτά. Εξού και το έγγραφό μας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε σχέση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι τεράστια και όχι μόνο για την Ευρώπη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο για τις στατιστικές υπηρεσίες. Δεύτερον, η σχέση με τους χρήστες. Εμείς ζητάμε από τις στατιστικές υπηρεσίες να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους χρήστες και υπό το φως των κινδύνων κατάχρησης των στατιστικών δεδομένων και κακής τους χρήσης γενικά. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες και σε χώρες που πρόσφατα αλλάξαν πολιτική ηγεσία, οι στατιστικές υπηρεσίες πιέζονται. Πιέζονται από κυβερνήσεις οι οποίες εμφανίζονται ότι είναι κατά τον ελίτ. Από ό,τι φαίνεται από τις έρευνες, τα στατιστικά δεδομένα θεωρούνται συχνά ένα από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ελίτ για να επιβάλλουν τις απόψεις τους πάνω στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί κάλλιστα και στην Ευρώπη, στο μέλλον, να αντιμετωπίσουμε πιέσεις προς τις στατιστικές υπηρεσίες να αλλάξουν την διακυβέρνηση και να ευθυγραμμιστούν περισσότερο προς τις επιθυμίες των κυβερνήσεων. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι η σχέση με τους χρήστες είναι κάτι που πρέπει να ενισχυθεί για να υποστηρίξουμε ακριβώς την ανεξαρτησία των στατιστικών υπηρεσιών. Τρίτη σύσταση. Με αυτές τις μεγάλες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, οι στατιστικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους και τους κατάλληλους πόρους, όχι μόνο οικονομικούς αλλά και ανθρώπινους. Δεν είναι εύκολο να προσλαμβάνει κανείς επιστήμονες που ασχολούνται με τα δεδομένα, γιατί στον ιδιωτικό τομέα ξέρετε ότι η κατάσταση είναι πιο ελκυστική, πληρώνουν πολύ περισσότερα. Όμως, είναι ζωτική σημασία στα δεδομένα και τα ψηφιακά δεδομένα για τις στατιστικές υπηρεσίες επόμενο σημείο. Η ηγετική θέση όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα. Όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικά τα στατιστικά δεδομένα για τη δημοκρατική συζήτηση. Και στην Ευρώπη γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν, δεν είναι σε θέση καν να διαβάσουν στατιστικά δεδομένα. Και μερικές φορές ακόμα και οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν την μεταφορά των στατιστικών δεδομένων με έναν τρόπο ιδιαίτερα χαλαρό. Γι' αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών Δεδομένων θα πρέπει να προσέξει περισσότερο αυτό το σημείο. Τώρα επιτρέψτε μου να περάσω περισσότερο σε βάθος στο έργο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Στατιστικών Δεδομένων. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι το στατιστικό αυτό σύστημα μπαίνει σε ένα νέο κύκλο αξιολόγησης μεταξύ ομοτήμων. Κάτι το οποίο βοηθάει τους ε, ανθρώπους που δουλεύουν στις στατιστικές υπηρεσίες και καταρτίζουν στατιστικές για να παρακολουθήσουν πιο καλά τον κώδικα δεοντολογίας που αποτελεί και το σημείο αναφοράς για την επαγγελματική ανεξαρτησία των ε, στατιστικών υπηρεσιών. Αρχίζει λοιπόν αυτή η αξιολόγηση. Εμείς ε, καταρτήσαμε κάποιες συστάσεις και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν, ελπίζουμε, γύρω στο 2022. Τρία χρόνια δουλειάς δηλαδή, για να καθοριστεί η μεθοδολογία ένας χρόνος πρώτα και δύο χρόνια για την αξιολόγηση αυτή καθε αυτή μεταξύ ομοτήμων. Και το 2020 θα παρέμβει βέβαια και ο συμβουλευτικός μας φορέας. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό που είναι πολιτικό είναι και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή δεδομένων. Γνωρίζουμε ότι χάρη στα μεγάλα δεδομένα, ε, πολλοί ιδιωτικοί φορείς που κατέχουν δεδομένα έχουν πλεονέκτημα για να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά σε σχέση με το δημόσιο τομέα. Εμείς λοιπόν ενθαρρύνουμε τις Εθνικές στρατιστικές Υπηρεσίες να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις με τον ιδιωτικό τομέα που κατέχει τέτοια δεδομένα, στην Ευρώπη για παράδειγμα, η κάθε χώρα θα έπρεπε να διαπραγματευτεί για τα δεδομένα αυτά με τον ιδιωτικό τομέα και να υπάρχει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση τελικά, ώστε αν μη τι άλλο οι στατιστικές υπηρεσίες να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους μέρος του πλούτου αυτού των δεδομένων που κατέχει ο ιδιωτικό τομέα. Και υπάρχει και μία σύσταση, που είναι βέβαια ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, και αυτό είναι ότι οι στατιστικέ υπηρεσίε θα έπρεπε να προσπαθήσουν και να φέρουν στην παραγωγή στατιστικών δεδομένων και αυτούς τους ιδιωτικούς φορείς που κατέχουν δεδομένα βάσει πάντα του κώδικα δεντολογίας και των ελάχιστων προδιαγραφών έτσι ώστε να διασφαλίσουμε συνολικά βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών δεδομένων, τόσο αυτών που παράγονται από το δημόσιο, όσο και αυτά που παράγονται από τον ιδιωτικό τομέα. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω και στις τελευταίες συστάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το μέλλον της διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Στατιστικών Δεδομένων. Θεωρητικά, ο ΕΣΚΑΠ, ο συμβουλευτικό Φορέας, πρέπει να καλύπτει την λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος συνολικά. Και η Eurostat πρέπει να ασχολείται με την ποιότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο. Όμως σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, σε λίγες, υπάρχουν και εθνικές αρχές οι οποίες έχουν τον ίδιο ρόλο. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ισχύει αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναπτυχθεί πολύ το σύστημα, στην Ιταλία όχι τόσο πολύ. τέλο πάντων, μόνο 6 από τις 28 χώρες διαθέτουν εθνικές αρχές. Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μας ελοχεύει κινδύνους, γιατί εμείς ως συμβουλευτικός φορέας δεν ε, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κανονισμό και να παρεύουμε στις εθνικές συνθήκες. Αλλά αν κανείς δεν το κάνει, τότε μπορεί να υπάρχει ανισορροπία. Εννοείται ότι η Eurostat κάνει πολύ και καλή δουλειά, αλλά η Eurostat υπάρχει γιατί ακριβώς ερμηνεύει τις συνθήκες, μπορούμε να πούμε. Συνεπώς εδώ έχουμε μια κρεμότητα και εξαιτία των κινδύνων που ελοχεύουν, όπως σας είπα πριν. Οπότε, ω συμβουλευτικό φορέα, σκοπεύουμε να οργανώσουμε φέτος μια συνάντηση με τους αντίστοιχού εθνικούς συμβουλευτικούς φορείς για να δούμε πώς μπορούμε παρετέρω να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών Δεδομένων. Το δεύτερο πολιτικό σημείο είναι το εξή. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, κάθε χώρα, κάθε κυβέρνηση, πιο σωστά, ενθαρρύνεται να εκδώσει μία δέσμευση εμπιστευτικότητας. Commitment of confidence. Ας πούμε να λένε εμείς θα στηρίξουμε ε, τον κώδικα διοντολογίας σε εθνικό επίπεδο περισσότερο. Λίγες χώρες όμως μέχρι τώρα έχουν εκδώσει τέτοιου είδους με μονομένες δεσμεύσεις. Ενώ Άλλε έχουν πει μα η νομοθεσία μας είναι ήδη ευθυγραμμισμένη και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με ένα τελευταίο σημείο που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας. Θα δούμε κατά πόσο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα προβληματιστούν όσον αφορά την διακυβέρνηση του Συμβουλευτικού Φορέα. Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτό στο μέλλον. Όπως επίσης και για αλλαγέ στις συνθήκες. Αυτό που εμείς έχουμε να συστήσουμε είναι ότι τελικά στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ΕΣΠΑΣ που είναι μια διοργανική προσπάθεια να γίνει κάποια έρευνα, μια μελέτη για να δούμε στο μέλλον τι ευκαιρίες μπορεί να υπάρχουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών Δεδομένων να αλλάξει τη διακυβέρνησή του. Δεν είναι κάτι καινούριο ότι εγώ προσωπικά είμαι υπέρ ενός ευρωπαϊκού συστήματος όπως αυτό που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά προς το παρόν καλό θα ήταν να εξεταστεί αυτό το θέμα, να μην υπάρχουν εκπλήξεις και έτσι το Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στα πλαίσια αυτά να αναλάβουν ηγετικό ρόλο για να υπάρξει αυτός ο προβληματισμός και αυτή η μελέτη για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζοβανίνη. Πολύ λογικές αυτές οι συστάσεις. Να ξεκινήσουμε με παρεμβάσεις των μελών. Ο κ. Γκέροντ για το ΕΛΚ ο πρώτος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την απουσία των συναδέλφων. Είναι κάτι συγκλονιστικό θα έλεγα. Μην θεωρείτε ότι είμαστε υπεύθυνοι, τους παρόντες γι' αυτό. Συστήνει στην και ζωντανή ότι η Eurostat και οι Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες πρέπει να διαμορφώσουν στρατηγική, σφαιρική, για τις σχέσεις με τους χρήστες. Όρια και δεδομένα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στα πλαίσια του εξαμήνου. Του SGBA τι προτείνει για να μπορούν να αξιολογήσουν σωστά την κατάσταση οι πολίτες και πώς ε, μπορεί να κρυθεί η θέση των διαφόρων χωρών όσον αφορά τα όρια για τα δεδομένα που έχουν καθοριστεί στο εξάμεινο. Απάντηση. Η βελτίωση της ευαισθησίας και της γνώσης του λαού για τα στατιστικά στοιχεία είναι με συστάσεις. Τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Όχι μόνο για διαμόρφωση πολιτικών, αλλά και για τις πολιτικές συζητήσεις και πολλές ψευδείς ειδήσει ε, διαβιβάζονται μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Όπως είπα, η ομάδα καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων ζήτησε από τις στατιστικές υπηρεσίες να ενεργοποιηθούν περισσότερο όταν γίνεται κακή χρήση των δεδομένων. Κατά παρελθόν, η βελτίωση των γνώσεων των πολιτών, το έργο αυτό, η εκπαίδευσή τους, και για τα στοιχεία που διαμορφώνουν την πολιτική ήταν κάτι που έκαναν οι εθνικές στατιστικές ε, ενώσεις. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι οι στατιστικές υπηρεσίες υπέχουν ιδιαίτερο καθήκον γι' αυτό σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης. Στην Ιταλία, όταν ήμουν πρόεδρος του Στατιστικού Ινστιτούτου, ε, φτιάξαμε ένα σχολείο με μαθήματα για τους δημοσιογράφους για την ανάλυση των στοιχείων. Ενθαρρύνουμε τι εθνικέ Στατιστικές υπηρεσίε να το κάνουν αυτό. Το Eurostat ήδη κάνει κάποια δουλειά σχετική, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι τη δημοκρατία. Κυρίω όταν είναι τόσο σημαντικά τα δεδομένα στο δημόσιο λόγο. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιε σχετικέ συστάσει, αλλά θα ήταν σημαντικό πιστεύω το Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί του πολίτε να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια, ούτω ώστε οι στατιστικές υπηρεσίες που είναι ανεξάρτητες από τις πολιτικές δυνάμεις να εκπαιδεύσουν τους πολίτες μέσω σχετικών προγραμμάτων για να βελτιωθούν οι γνώσει όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία. Μην ότι μετά τη χρηματοστατική κρίση οι κεντρικές τράπεζες ξεκίνησαν σε μαζική κλίμακα προγράμματα για την ενημέρωση του λαού για τα χρηματοπιστωτικά, για να αποφευθούν τα προβλήματα που οδήγησαν μεταξύ άλλων στη χρηματοπιστωτική κρίση. Παρόμοια προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί και για την εκμάθηση των στατιστικών στοιχείων με την υποστήριξη των εθνικών ε, φορέων που παράγουν τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Υπερβάμς Περέζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον καλεσμένο μας. Στο ΕΣΚΑΠ αυτό το πνεύμα θέλαμε να πριτανεύει. Είπατε ότι 6 με 7, αν μετρήσουμε τον μεν Βασίλειο, όχι, χώρες, είπατε, έχουν ανεξάρτητες στατιστικές υπηρεσίες ή φορείς που εποπτεύουν σε εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Και αναφερθήκατε στους κινδύνους που ελοχεύουν όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία που μπορούν να χειραγωγούνται από κάποια συμφέροντα. Η νομοθεσία είπατε ότι δεν επιτρέπει στην ΕΣΓΑΜ να παίξει αποφασιστικό ρόλο στον έλεγχο της χρήσεως των στατιστικών στοιχείων και πώς εφαρμόζει η ειδική νομοθεσία στα κράτη-μέλη, είπατε ότι θα το επεξεργαστείτε το θέμα. Μπορείτε να μας αποκαλύψετε ποιο, ποιοι δρόμοι διαφαίνονται για την Ένωση για να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Παρομοίως. Για την ευρωπαϊκή διαχείριση του θέματος, τη δίκηση, ποιο ρόλο βλέπετε ότι μπορεί να παίξει η Εθνική Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία στα πλαίσια της, α, του θεματολογίου του ΟΗΕ για το 2030 που θα εκδοθεί αύριο. Μετά, για να μπούμε στην ουσία. Συλλογή πληροφοριών από πλευράς Eurostat. Επεξεργαζόμαθα πολύ τα θέματα της φοροδιαφυγής και των διαφορών μεταξύ πολιτικών, του policy gap, το φορολογικό κόστος που απορρέει από τα μέτρα που, δημιουργούν, που εφαρμόζουν κάτι μέλη και δημιουργούν ε, διάφορες δυνατότητες μη καταβολής των φόρων. Και αυτό είναι μια πηγή αποξήρανσης το υπήν των δημοσίων εσόδων. Έχετε ιδέες από αυτόν. Η επικαιρότητα προωθεί αυτό το θέμα και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες επεξεργαζόμεθα το θέμα αυτό, εντοπίζουμε υπό την ηγεσία του Ρίτσαρντ Μέρφυ το policy gap που υπάρχει. Συναρτήσει των συμπεριφορών, συμπεριφορών των διαφόρων κυβερνήσεων. Και βάσει των δεδομένων ε, του 2015 η απώλεια ανέρχεται σε 825 δις ευρώ. Έχετε συστάσεις Έχετε επιθυμίες όσον αφορά το πόσο χρησιμοποιούνται τα στατιστικά στοιχεία από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι εμεί καταρτίζουμε ένα ευχολόγιο του ΣΥΠΗΝ ε, που θα απευθυνθεί προς την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Η δυνατότητα δημιουργίας εθνικών φορέων παρομοίων με την ΕΣΓΑΠ, που θα είναι ανεξάρτητοι φορείς, οι οποίοι φορείς αυτοί θα ελέγχουν τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες είναι μια δυνατότητα για καλύτερη κάλυψη του συστήματος. Μια άλλη δυνατότητα είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι η SGAB έχει δικαίωμα να μπορεί να επιληφθεί του θέματος και να εξετάζει τις καταστάσεις στα διάφορα κατημέλη. Τι εννοώ. Παραδείγματο χάρη, στην εξέταση των έλεγχων μοτίμων που ήδη λαμβάνει η χώρα υπήρχαν κενά. Εντοπίστηκαν κενά σε διάφορες χώρες. Ανάλογα με την ερμηνεία του ρόλου της ΕΣΓΑΠ μέχρι τώρα, στην έκθεσή μας δεν μας επιτρέπεται να αναφέρουμε συγκεκριμένες εθνικές περιπτώσεις και το σύστημα στο σύνολό του. Δεν το αναφέρει ρητά ο κανονισμός, άρα είναι θέμα ερμηνείας και θέμα πόρων βέβαια. Μη λησμονούμε ότι στην ΕΣΓΑΠ δωρεάν παρέχουμε υπηρεσίες, η γραμματεία είναι πάρα πολύ μικρή. Αν το Κοινοβούλιο λοιπόν θέλει εμείς να μπούμε εις βάθος εξετάζοντας τις εθνικές καταστάσεις πρέπει να επαναξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας μας και πόσο θα μας υποστηρίζει το έργο μας στο Eurostat. Δεν έχω ακόμα κάποια λύση. Θα ακολουθήσουν συζητήσεις στους επόμενους μήνες και αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει να διευκρινίσουμε τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων επιλογών. Και μετά ενδεχομένω θα υποβληθεί η κατάλληλη πρόταση. Για το δεύτερο ερώτημά σας για τη νέα ατζέντα, για τις νέες δραστηριότητε μάλλον, που ίσως θέλει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε το θεματολόγιο του 2030, του 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη να συμπεριληφθεί στις δραστηριότητε της, είναι ένα άλλο θέμα. Θα δούμε τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτό. Α, υπάρχει και μία δυνατότητα βέβαια. Μία από τι δυνατότητε είναι να αλλάχθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο καλύπτοντας και άλλους τομείς ή ακολουθώντας πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανάλυση περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική. Εν αυτή η περιπτώση είναι απαραίτητο να καταβληθεί προσπάθεια επιτάχυνσης της παραγωγής κάποιων στοιχείων. Παραδείγματο χάρη, στοιχεία που αφορούν το κοινωνικό τομέα, ούτω ώστε τα δεδομένα να ευθυγραμμιστούν με τα οικονομικά στοιχεία. Μη ότι όταν συζητούμε συστάσεις αναχώρα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία έχουμε στοιχεία για το ΑΕΠ που είναι επικαιροποιημένα μέχρι το τελευταίο τρίμηνο. Ενώ για την διανομή του εισοδήματος, κατανομή εισοδήματος, έχουμε ε, στοιχεία που χρονολογούνται προ δύο ετών. Και έτσι δημιουργείται έλλειψη ισορροπίας, ανισορροπία. Το ίδιο ισχύει και για τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Νομίζω, συνεπώς, ότι αυτή η Επιτροπή θα μπορούσε πραγματικά να αξιολογήσει ενδελεχώς αυτά τα ζητήματα, διότι πρόκειται περί της ποιότητας των αποφασιών σας. Αυτό είναι ένα και μόνο παράδειγμα του πώς το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα συγγνώμη, μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία του για να υποστηρίζει και εσά τη διαδικασία ως αποφάσεων. Όσον αφορά τα θέματα τα δημοσιονομικά, τα φορολογικά, και αυτά τα κενά, τα φορολογικά που αναφέρατε. Διαφορετικό θέμα είναι αυτό. Αυτό απαιτεί πολλούς υπολογισμούς, υποθέσεις, μοντέλα, εκτιμήσεις. Το Eurostat μπορεί να παράσχει βοήθεια. Δεν είναι αποκλειστικά στατιστικό θέμα και εγχείρημα και γι' αυτό μέχρι τώρα οι στατιστικές υπηρεσίες δεν έχουν εμπλακεί αλλά είναι σημαντικότατο ζήτημα και ο Πρόεδρος προανέφερε ότι θα ψηφίσετε το, για το καθάριστο χώριο προϊόν που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο κίνδυνος να αναπτύσσεται η οικονομία η γκρίζα λόγω αυτών των καταστάσεων είναι πραγματικός. Γι' αυτό ε, το Eurostat θα μπορούσε να βοηθήσει στην ε, αξιολόγηση που ίσως ζητήσετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Σύντομη η συζήτηση. Ε, η κυρία Περέζε, εκτό μικροφώνου, δεν την ακούν οι διερμήνεις. Α, συγγνώμη. Είπατε κάτι για την Κομισιόν, λέει και ο Τζοβανίνη. Η θέση, οι ευθύνε της Eurostat εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι κάτι εύκολο να καθοριστεί, διότι είναι οριζοντίου χαρακτήρα τα στατιστικά στοιχεία. Από καιρού καιρών οι ευθύνε μετακινούνται και πάνε από έναν επίτροπο σε άλλον. Εγώ δεν έχω κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως ότι στην αξιολόγηση που πρέπει, όσον αφορά το Commitment of Confidence αναγνωρίσαμε ότι πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριζε και σεβόταν το έργο του Eurostat. Αυτό που δεν θα συνέστηνα θα ήταν να επιστρέψουμε στην παλιά κατάσταση, όπου τα στατιστικά στοιχεία ανήκαν μαζί με το φορολογικό έλεγχο, το δημοσιονομικό έλεγχο και τις άλλες διοικητικές ευθύνες. Τώρα τα στατιστικά στοιχεία στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πηγαίνουν μαζί με την ενία αγορά. Αυτή είναι μια επιλογή, αλλά είναι πραγματικά απαραίτητο όποιο είναι υπεύθυνο για τα στατιστικά στοιχεία να σεβαστεί το, το θέμα της εμπιστευτικότητα, το commitment of confidence και ετοιμάσει και νέα τέτοια δέσμευση περί εμπιστευτικότητα. Έτσι θα εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και του Eurostat και άλλων υπηρεσιών όταν παράγουν ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια συζήτηση ε, σε μικρό, σε στενό κύκλο, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο καθηγητής Τζοβανίνη πάντα διασύνδε σαφώς τα διάφορα τεχνικά ζητήματα, υπογράμμιζε τις σχετικές πολιτικές και προκλήσεις, πάντα ήταν ξεκάθαρος, ευχαριστώ για τη μεθοδό σας. Εκτιμούμε τον τρόπο παρουσίασης Ευχαριστούμε για τις συστάσεις, τις πληροφορίες και για τα προβλήματα που εντοπίσατε και ελπίζω ότι το επόμενο κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε την σκητάλη στο επόμενο κοινοβούλιο και εμείς που θα είμαστε παρόντες στο επόμενο κοινοβούλιο να συνεχίσουμε τον επικοδομητικό διάλογο και τη συνεργασία με την ΕΣΚΑΠ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Ζωβανίνη, καθηγητή Τζοβανίνη. Ευχαριστώ την απερχόμενη Επιτροπή ΕΚΟΝ για την υποστήριξή τη. Έχει δώσει στην ΕΣΚΑΠ με την πάρο των ετών την προσοχή που αξίζει την ΕΣΚΑΠ. Ευχαριστούμε τα μέλη για την προσοχή που έδωσαν στα στατιστικά θέματα και ελπίζω ότι το νέο κοινοβούλιο θα κάνει τουλάχιστον τα ίδια, θα έχει τουλάχιστον την ίδια στάση και όπως είπατε ενδεχομένω θα δοθεί μεγαλύτερη ακόμα προσοχή, διότι αυτά τα θέματα είναι σημαντικά από πλευρά πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Διακόπτουμε σύντομα, διότι μετά έχουμε κοινή συνεδρίαση οίκων και budget για την μεταρρύθμιση του ESM.